να ε, προβλεφτούν μόνο εάν υπάρχει η ομόφωνη άποψη των ε, κρατών μελών. Κλείνει η συζήτηση. Αύριο την Τρίτη είναι η συζήτηση. Η ψηφορία με συγχωρείτε. Πάμε τώρα στην ε, έκθεση Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση που συζητάμε αφορά κυρίως ε, τα διορθωτικά ε, ταμεία και τι ε, δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση. Η οικονομική κρίση έχει ε, επιβάλει αυστηρότερου ε, νόμου και έχει επιβάλει περικοπές χωρίς καμία απολύτω διαφοροποίηση ανάμεσα επενδύσει και τα πάγια έξοδα. Αποτέλεσμα αυτού περιορίστηκαν σχεδόν πλήρω οι πολιτικέ που έχουν ω στόχο την οικονομία και την ανάπτυξη. Αυτό βέβαια είχε συνέπειες στην πολιτική συνοχή και οι ε, δαπάνες για τις επενδύσεις είναι όμως απαραίτητες για να ξεπεραστούν ε, οι διάφορες ανισότητες που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση καλείται να εφαρμόσει την ευρωπαϊκή πολιτική αλλά έχει δυσκολίες. Της είναι δύσκολο να εφαρμόσει όλα αυτά τα προγράμματα τα στοιχεία σχετικά ε, με τις περικοπές και τη διαφορά ανάμεσα στις ισχυρές και τις αδύναμες ε, πολιτικές δείχνουν ότι έχουμε όλο και λιγότερη συνοχή. Υπάρχουν λοιπόν τρεις προτάσεις για να υπάρχει ισορροπία, να εξισορροπηθούν οι επενδύσεις με τις απαιτήσει για ε, λιτότητα και περικοπές. Να πούμε λοιπόν το εξή. Η πρώτη παραδοχή είναι, η πρώτη πρόταση είναι ότι οι δαπάνες θα πρέπει να ξεκινούν από το έλλειμμα και την αντιμετώπιση του. Οι δαπάνες αυτές έχουν ως στόχο να αντιμετωπιστούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020, κυρίως όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή όμως δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και έτσι λοιπόν από τη μια ε, περικόπτουν οι δαπάνε, από την άλλη όμως υπάρχουν και κυρώσεις γιατί δεν γίνονται οι δαπάνε. Η δεύτερη πρόταση είναι ότι στον υπολογισμό, εν πάση περιπτώσει, των ε, δαπανών και του βάρους που συνδέεται με τις επενδύσεις, αυτό να συνδέεται με ε, τους φόρους, με την επιβολή των φόρων. Ας μην ξεχνάμε ότι και αυτοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στον ορισμό του ελλείμματος. Και η τρίτη πρόταση είναι στον προϋπολογισμό, στην αρχή του, ε, του προγραμματισμού, να εντάσσεται το συνολικό ποσό των ε, κοινοτικών κονδυλίων και η εθνική συμμετοχή να αναφέρεται στους επόμενους ε, προϋπολογισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να επιτύχουμε μια εξορρόπηση με τα προηγούμενα προηγούμενα έτη και με τις επενδύσεις που είναι απαραίτητες. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι με την έκθεση αυτή θέλουμε να απευθυνθούμε στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις οι οποίε έχουν διατυπωθεί και στο πλαίσιο του πακέτου συνοχής. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό αναφέρεται και στην εντολή που έδωσε η Επιτροπή περιφερειακών υποθέσεων στους ε, εισηγητές. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι εργαζόμεθα όλοι συνεπείς. Και κατά τα άλλα ε, η έκθεση αυτή έφτασε εδώ στην Ολομέλεια σχεδόν με απόλυτη ομοφωνία με 40 πέρ και μόνο δύο αποχές. Και επιπλέον προστίθεται και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Προπολογισμών και η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Εργασίας. Η έκθεση αυτή νομίζω ότι σχετίζεται άμεσα και με τη συζήτηση που ξεκίνησε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, σχετικά με την ε, εισαγωγή χρυσών κανόνων στη φορολογική πολιτική. Να έχουμε μια Ευρώπη ε, που να είναι ευφυής, ευαίσθητη μέχρι το 2020. Έτσι λοιπόν κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προάγει την απασχόληση, να προάγει την ανάπτυξη των υποδομών, να δώσει ανάκαμψη στην οικονομία γιατί αλλιώς δεν είναι δυνατόν να επιληθούν οι, ε, τα προβλήματα εκείνα τα οποία έχουν προκληθεί. Εγώ λοιπόν έχοντας όλα αυτά κατά νου εύχομαι το Κοινοβούλιο να μπορεί με ευνοϊκή ψήφο να καταδείξει ότι και αυτό δραστηριοποιείται και έχει σαφή γνώση του ρόλου του ως ε, νομοθέτης δεν αφήνει ε, μικρά συμφέροντα να επικρατούν και να επικρατούν εθνικιστικές απόψεις. Πάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye ε, και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θαυμάσια η έκθεση της Αντέλεφου κυρίας Ματσόνη γιατί προσφέρει συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την απαραίτητη ευελιξία σε σχέση με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες προτεραιότητες που αφορούν στις επενδύσεις, στις δημόσιες επενδύσεις και νομίζω πρέπει να σας επενθυμίσω ότι περίπου το 60% των επενδύσεων γίνεται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξάλλου θα πρέπει από το Σύμφωνο Σταθερότητας να εξαιρείται το ποσοστό της εθνικής συγχρηματοδότησης. Μιλάμε για στρατηγικές δαπάνες καθοριστικής σημασία για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Μιλάμε για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της εργασίας. Νομίζω πρέπει να το επενθυμίσουμε ότι το Σύμφωνο λέει ναι στη σταθερότητα αλλά και στην ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να πεθάνουμε από τη λιτότητα. Ευχαριστούμε την κυρία Αντζελίλη. Ο κύριος Ταμάζη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε ε, Επίτροπε. Θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, συναδέλφους για αυτή την εξαίρετη έκθεση. Ε, η πολιτική συνοχή είναι πολύ σημαντική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς υπάρχουν ε, μεταξύ του 2014 και το 2020 πολύ λίγα μέσα ε, πολιτικής συνοχής και αυτό το εξέθεσε πολύ καλά η κυρία Ματσόνη. Συγκεκριμένα οι κανόνες, οι μακροοικονομικές προϋποθέσεις είναι μια πολύ κακή πρόταση, είναι πολύ μεγάλη ευελιξία που δίνουν. Η πολιτική συνοχή λοιπόν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, όπως την παρουσιάζει η κυρία ε, Ματσόνη. Να μην υπάρχει έλλειψη δηλαδή μέσων. Να μπορούν τα κράτη-μέλη να υποστηρίζουν ε, τα μέτρα της συνοχής. Ευχαριστώ πολύ και υποστηρίζω την έκθεση. Ευχαριστούμε τον κύριο Μπάτζη. Δίνω το λόγο στον κύριο Γκάουιν. Εκτός μικροφώνου ο μιλητής. Κύριος Γκάλαχερ, εκτός μικροφώνου. Του region has been greatly affected by rising unemployment levels as a result of the economic recession. Despite this... Παρά το γεγονός ότι η, η περιοχή ήταν πολύ πιο αναπτυγμένη εξαιτία ε, των επιπέδων που χρησιμοποιήθηκαν ε, ΑΕΠ ε, κατά κεφαλήν. Η περιοχή αυτή πήρε 100 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα λάβει στοιχεία σχετικά με τη μείωση στα κονδύλια. Θεωρείται ότι η περιοχή αυτή ε, μέσα από το Leader ε, προσπάθησε να χρησιμοποιήσει κονδύλια μέσα από τη συγχρηματοδότηση. Thank you very much. I give... Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χρυσόγελος έχει το λόγο. αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα. Yes. Okay. Ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο γιατί πραγματικά μιλάει για την ουσία του προβλήματος. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα δημοσιονομικά προβλήματα αλλά απ' την άλλη η κρίση και η πολιτική λιτότητα έχουν οδηγήσει σε χειρότερα προβλήματα. Α δούμε για παράδειγμα την Ελλάδα, έχει καταρρεύσει η οικονομία τη, έχει τεράστια προβλήματα ανεργία, έχει επιδεινωθεί το χρέο και διαλύεται η κοινωνική τη συνοχή. Τι πρέπει να κάνουμε για να καλύψουμε τη μείωση των δαπανών από το δημόσιο θα έπρεπε να αυξηθούν οι δαπάνες από τις περιφέρειες να ενισχυθεί η οικονομία αλλά ακριβώς αυτές οι περιφέρειες που έχουν περισσότερο ανάγκη από επενδύσεις αυτές αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα γιατί χάνουν και πόρους από τον κρατικό προπολογισμό και ιδίους πόρους και αντιμετωπίζουν προβλήματα και με το προσωπικό που χάνεται. άρα οι στόχοι της ευρώπης 2020 είναι πιθανό να μην επιτευχθούν πώς θα γίνει; πρέπει λοιπόν το ταμείο συνοχής και τα άλλα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να ενισχύσουν τόσο τις περιφέρειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και την κοινωνική οικονομία να υπάρξει ευελιξία στα προγράμματα να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων και οι ίδιες οι περιφέρειες να αυξήσουν την ικανότητά τους να απορροφούν προγράμματα γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που δεν μας βγάζει σε συνοχή αλλά εντείνει τις ανισότητες και τις διακρίσεις μεταξύ των περιφερειών και αυτό το βλέπουμε όχι μεταξύ των περιφερειών στην ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό κάθε χώρας και στο εσωτερικό κάθε περιφέρειας. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή, η οποία υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η δραστηριοποίηση της κάθε περιφερειακής πολιτικής για την πολιτική συνοχή. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω τις προτερότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις συνδυάσουμε με τους περιφερειακούς και τοπικούς στόχους. Αυτό στο κάτω-κάτω είναι ο ρόλος της πολιτικής συνοχής οι τοπικές ομάδες μπορούν να βοηθήσουν πολύ. Πρέπει να φροντίσουμε όμως να έχουμε καλή ισορροπία από τη μια μεριά τα μέτρα, τα διορθωτικά εξυγίανσης των δημοσιονομικών και από την άλλη μεριά όμως να έχουμε την ανάπτυξη. Αλλιώ δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη σε πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Κυρία Τόμαζιτς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έρχομαι από την Κροατία. Οι περιφερειακές μας δομές δυσκολεύονται πάρα πολύ με την βιωσιμότητα και θέλω αυτό να σας το υπογραμμίσω εδώ. Δεν πρέπει να επιμένουμε να εφαρμόζουμε ένα και το ίδιο μοντέλο σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί κάθε δομή δεν έχει τον ίδιο βαθμό αποκέντρωσης, για παράδειγμα. Συμφωνώ ότι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες πρέπει να θαρρυνθούν και να πετύχουν υψηλότερη ανάπτυξη, αλλά δεν θα πρέπει από την άλλη μεριά πιο πλούσιες περιοχές να νιώθουν ότι υπάρχει κατάχρηση σε βάρος τους από τους πιο φτωχούς τα διάφορα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Τα πλούσια κράτη-μέλη μπορούν να μας προσφέρουν περισσότερα από ότι απλώς χρήματα. Μπορούν να μας δώσουν συμβουλές, να μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε καλά τις μεταρρυθμίσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα το σύστημά μας να είναι πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε λέει κυρία Σουίκα. Ξέρουμε ότι έχουμε λιτότητα σε πολλές χώρες, περικοπές από την κεντρική κυβέρνηση. Από την άλλη μεριά βέβαια οι ίδιες χώρες που έχουν αυτά τα προβλήματα πρέπει να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες. Οι περιφερειακές κυβερνήσεις πρέπει να προσπαθήσουν συνεπώς να κάνουν ευθύς επενδύσεις, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα όσο γίνεται καλύτερα. Η πρόταση αυτή έχει στηριχθεί με μεγάλη πλειοψηφία. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένα μέτρα, την απασχόληση και να μπορέσουμε με ανταγωνιστικό τρόπο να έχουμε ανάπτυξη. Οι δημόσιες δαπάνες δεν θα πρέπει να υποφέρουν όπως γίνεται σήμερα σε πολλές χώρες μέλη. Θέλω λοιπόν να στηρίξω αυτούς που θέλουν να αλλάξουν οι κανόνες και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στην χρήση των διαφορετικών κονδυλίων ώστε έτσι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε πιο γρήγορα τα προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι πολύ σημαντικό για την Κροατία που τώρα αρχίζει να χρησιμοποιεί τέτοια κονδύλια. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Φερέιρα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η έκθεση αυτή αναγνωρίζει μια σαφή τάση που είναι η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όμως έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με την ολοκλήρωση, με τις κοινέ πολιτικές. Πολιτικές οι οποίες όμως έχουν έναν φιλελεύθερο τόνο, άρα ενισχύουν τις διαφορές και τις ανισότητες. Είναι μια δυναμική η οποία χωρίς κανένα πρόβλημα προχωράει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τροποποίηση στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της κάθε περιφέρειας στην ανάπτυξη και το δικαίωμά της να χρησιμοποιήσει το ίδιο το δικό της δυναμικό. Αύξηση των κονδυλίων για την οικονομική και κοινωνική συνοχή και όχι αποδυναμωσή τους όπως προβλέπεται με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης πρέπει να αποφύγουμε τις απώλειες κονδυλίων και να σταματήσουν οι μακροοικονομικές ε, απαράδεκτες προϋποθέσεις. Πρόεδρος. κύριος Κέλλη. Ως μέλος ε, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, θα ήθελα να επενέσω την εισηγήτρια. Τον τελευταίο καιρό έχουμε προχωρήσει από την απλούστευση στην ευελιξία. Και εάν ε, μπορούμε λοιπόν να ε, επιδιώξουμε αυτούς τους στόχους ε, θα σημειώσουμε μεγάλη πρόοδο και τα χρήματα θα δαπανώνται προς όφελος των πολιτών το ΑΕΠ αναφέρθηκε αυτό ε, δεν είναι το βέλτιστο μοντέλο για να το χρησιμοποιούμε ως ε, σημείο αναφοράς. Αυτό αναφέρθηκε από όλου. Αυτό που έχει σημασία είναι να γίνεται το καλύτερο για την ε, τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σάντσες Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν είναι κάτι ουδέτερο. Η Ευρώπη από το 2050 έχει επενδύσει 350 εκατομμύρια για την ανάπτυξη των περιφερειών. Τα κονδύλια αυτά αποτελούν μοχλό για την ενίσχυση των δημοσιονομικών ε, των ε, περιφερειών που πρέπει να προσθέσουν κάθε φορά χρήματα. Από την άλλη μεριά, εξαιτία των περιορισμών, δυσκολεύονται να προσθέσουν τα χρήματα αυτά οι περιφέρειες και το αποτέλεσμα είναι να μην γίνονται καθόλου επενδύσεις. Τελήματα είναι υπεύθυνα. Ο καλύτερος τρόπος για να δαπανάμε πρέπει να είναι η αρχή μα για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι χώρε και για τι περιφέρειες. Χρειάζεται ευελιξία, αλλά οι περιφέρειες πρέπει να τηρούν τι υποχρώσεις του απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρούν το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα για τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Τότε μόνο η ανάπτυξη μπορεί να προχωρήσει σε στέρεες βάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κυρία Μπόρτζα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η, Επιτροπή, η πολιτική συνοχή είναι το πιο σημαντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην μάχη του κατά της ύφεσης. Όμως οι δημοσιονομικοί περιορισμοί μπορεί να καταργήσουν τις θετικές επιπτώσεις της, Επιτροπής, της ε, πολιτικής συνοχής. Η λιτότητα σε εθνικό επίπεδο και η δυσκολία χρηματοδότησης των τοπικών προγραμμάτων θα έχουν σημαντικό και επίπτωση στις δυνατότητες καλής χρήσης των διαρθρωτικών ε, ταμείων. Το... Αυτό ο ε, ε, αυτές οι μονάδες, οι τοπικές και περιφερειακές που είναι πιο ευαίσθητες, αυτές θα πληγούν περισσότερο. Είναι λοιπόν σημαντικό τώρα να μιλήσουμε για εξαιρέσεις. Είναι το βήμα προς την κατάλληλη κατεύθυνση, διότι μιλάμε για πόρους που έχουν στόχο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Επίτροπη. Στην χώρα μου προσπαθούμε να μεταφέρουμε μέτσα, μέτρα συνοχής έτσι ώστε να μπορέσουμε να, ε, να έχουμε ε, πρόοδο. Για παράδειγμα έχουμε γέφυρες οι οποίες ε, χτίζονται μεταξύ της Πρατισφλάβα και άλλων πόλων. Υπάρχει σημαντικό... Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν σημαντική μεταφορά κονδυλίων, όμως αυτό οδήγησε σε μείωση κατά 10% των επενδύσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, για να επιτύχουμε μια εναρμονισμένη εξέλιξη των περιοχών, θα πρέπει να υπάρχει ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στις τοπικές ομάδες να έχουν στρατηγικές για βιώσιμη ανάπτυξη. Η εφαρμογή ενός τέτοιου μέσου θα βελτιώσει την απλούστευση των κανόνων και θα αυξήσει την ευελιξία σε επίπεδο σχεδιασμού και χορήγησης ε, κονδυλίων. Σε μια περίοδο λοιπόν ε, στασιμότητας ε, θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην βελτίωση της προσβασιμότητας στα ευρωπαϊκά ταμεία. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Δαμανάκη, την Επίτροπο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, αλλά επίσης ε, συμμεριζόμαστε και τις ανησυχίες ε, που εκφράζονται στην έκθεση της κυρίας Ματζόνη. Η οικονομική κρίση πραγματικά ε, αποκάλυψε ε, τη διαδικασία συνοχής ότι η διαδικασία συνοχής έχει προβλήματα εξαιτίας της αύξησης των ανισοτήτων, ειδικότερα σε τοπικό επίπεδο. Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι οι βασικοί παίχτες που θα βελτιώσουν την κατάσταση στην Ευρώπη μετά από αυτή την κρίση. Το πάνω από 46% των ε, δαπανών για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών μελών δόθηκε ε, από υποεθνικές αρχές, ε, δηλαδή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι κυβερνήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έκαναν πολύ σημαντικές δημόσιες επενδύσεις. Το 2012 περίπου το 60% των δημοσίων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έγινε από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η οικονομική κρίση έχει μειώσει τους πόρους για τις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Αυτό είναι αλήθεια. οι δαπάνες σε δημόσιο επίπεδο έχουν συρρικτωθεί δραματικά. Το 2011 οι δημόσιες επενδύσεις έπεσαν στο 2,1 στα επίπεδα δηλαδή του 1997. Σε πραγματικούς όρους, ε, οι δημόσιες επενδύσεις από τοπικούς και περιφερειακούς ε, τομείς έπεσαν σε, στο κατά 5,7% το 10, 6,7% το, 12, το 11 και το 2012 ακόμα περισσότερο. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Πολλά κράτη-μέλη έχουν, έχουν δηλώσει ότι έχουν πρόβλημα με τη συγχρηματοδότηση των ε, έργων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι δείχνει ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει σοβαρά την ικανότητα των περιφερειακών και τοπικών αρχών να κάνουν δημόσιες δαπάνες, οι οποίες είναι κρίσιμες έτσι ώστε να διατηρηθεί η προοπτική για ανάπτυξη στο μέλλον. Η Κομισιόν έχει προτείνει μια σειρά μέτρα για να βελτιώσει την δημοσιονομική διαχείριση αυτών των πόρων. Καταρχάς, έχουμε προτείνει μεγαλύτερα ποσοστά συγχρηματοδότησης ε, μέσα από την υποστήριξη στην τρέχουσα περίοδο και στο μέλλον. Δεύτερον, η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί την ε, πιο αποτελεσματική χρήση των ε, πόρων. Ειδικότερα θα πρέπει θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην στρατηγική Ευρώπη 2020 να πλουστευτούν οι διαδικασίες και να ενθαρρύνουμε τη χρήση των ευρωπαϊκών ε, μέτρων. Επίσης, η, πολιτική συνοχή θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις μακροοικονομικές ε, προοπτικές ε, του ευρωπαϊκού εξαμήνου έτσι θα έχουμε πιο στενούς δεσμούς μεταξύ συνοχής και μακροοικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό έγινε μέσα από, τις, ε, μέσα από τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Ταυτόχρονα η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι θα επιτρέπει, υπό όρους φυσικά, προσωρινές παρεκκλήσεις από τις απεπτήσεις ε, του προληπτικού βραχίωνα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έτσι ώστε η εθνική συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να εξυπηρετηθεί. Θα πρέπει, ε, πρόσφατα επίσης η Κομισιόν ε, εξήγησε τις λεπτομέρειες αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει η συζήτηση. Αύριο, 3η, ε, 8 Οκτωβρίου στις 12 είναι η ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στην έκθεση Έλλης. Δίνω το λόγο στον κύριο James Ellis.